Uh, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας μετά από ένα καλό γεύμα, ελπίζω. Θα μιλήσουμε ε, για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, όπως κάναμε και προηγουμένως, αλλά ειδικά σήμερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως πολιτικοί ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι μικρομισές επιχειρήσεις και μιλούμε πάντοτε για αυτές ε, σε όλες τις χώρες πριν από τις εκλογές, αλλά νομίζω ότι ο τομέας είναι πραγματικά σημαντικός ε, για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, εφόσον έχουμε καθυστερήσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θα ακολουθήσουμε το πρόγραμμα. Έχουμε τρεις ομιλητές προσκεκλημένους ε, Χαιρετίζω τον καθηγητή Άλλερς, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής μιας μικρομεσαίας γερμανικής επιχείρησης ε, και αντιπροσωπεύει επίσης και την Ένωση στην Ευρωπαϊκή, τον κύριο Γκούς, ο οποίος είναι Πληρωματικός εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και τον κύριο Τοκάρσκι, επικεφαλής της ε, ε, Γενικής Διεύθυνσης Επιχείρησης και Βιομηχανίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνο της μονάδας. Νομίζω ότι θα έχει 10 λεπτά ο καθένας από εσά τους τρεις και μετά θα έχουμε χρόνο για έρωτα απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω κυρίες και κύριοι σήμερα για αυτήν ε, την ακρόαση. Ονομάζομαι Άλλερς και αντιπροσωπεύω την ε, SD εκ μέρου ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αλυσίδα εφοδιασμού και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Γερμανία που είναι, δραστηριοποιούνται στην αεροναυτική και το διάστημα. Ξέρω λοιπόν από τις επιχειρήσεις ότι, που ενδιαφέρονται για την τυποποίηση και θέλουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας και ε, ενδιαφέρονται για την ASD, Aerospace and Defense. Θέλουμε να δούμε πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται ε, στην αλυσίδα εφοδιασμού και στην ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αργότερα επίσης ε, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτα απ' όλα αν μιλήσουμε για την Ευρώπη μπορούμε να πούμε ότι δύο από τις τρεις θέσεις εργασίας ε, στον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από την άλλη πλευρά πάνω από, το, ε, από τη μισή προστιθέμενη αξία δημιουργείται από αυτές τις επιχειρήσεις. Εξαρτώμεθα λοιπόν από αυτές ε, τις βιομηχανίες των μικρομεσαίων αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε μεγάλη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών σε σχέση με καινοτόμες νέες τεχνολογίες και ότι είναι απαραίτητο για έρευνα και ανάπτυξη και εφαρμογές σχετικά με τον τομέα αυτό. Από αριθμούς αυτό σημαίνει ότι 80% των προμηθευτών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τώρα ε, μπορείτε έτσι να δείτε περίπου ποια είναι η σημασία του τομέα αυτού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αν μιλήσουμε για τεχνογνωσία και για καινοτομία, τότε θα βρείτε ότι οι περισσότερες από τις προτάσεις που βρίσκεται στις νέες τεχνολογίες, στις νέες προϊόντα στην αγορά σχετίζονται επίσης με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τεχνογνωσία εμπειρογνωμοσύνη που περιλαμβάνεται σε μεγάλα έργα και προγράμματα σχετίζονται με επιτεύξεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνεπώς, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έρευνα, τεχνολογία και ανάπτυξη με τέτοια προγράμματα, ούτως ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν με την δουλειά τους και να περιλάβουν τις καινοτομίες αυτές στα νέα προϊόντα και εφαρμογές. Δεν θα μιλήσω για την ευελιξία και τα κίνητρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι θέλουν να επιβιώσουν στην αγορά και με την έρευνα και τεχνολογία είναι σημαντική για αυτούς το, η έρευνα και τεχνολογία, αλλιώ δεν μπορούν να επιβιώσουν στην αγορά. Όταν μιλήσουμε για την σχέση μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μεγάλων συστημικών επιχειρήσεων, τους, αυτούς τους κατασκευαστές του εξοπλισμού, βλέπουμε ότι ενδιαφέρονται ε, για την ολοκλήρωση των μεγάλων συστημάτων, υποσυστημάτων, για τα νέα αεροσκάφη, ε, για τα σκάφη του διαστήματος και για τα ελικόπτερα. Και αυτό μας βάζει εμάς τις μικρομεσαίες ε, σε θέση να θέλουμε να μάθουμε τι συμβαίνει με τις μεγάλες εταιρείες διότι θα πρέπει να έχουμε πελάτες, θα πρέπει... Δεν πρέπει να, πρέπει να κάνουμε κάτι επειδή αξίζει και επειδή μπορούμε να έχουμε το μερίδιό μας στην αγορά αυτή για το μέλλον. Δυστυχώς το μερίδιο της αγοράς στο μέλλον σημαίνει στην αεροναυτική και στον τομέα του διαστήματος ότι πρέπει να περιμένουμε 5 με 10 χρόνια μέχρι ότου να μπορούμε να σκεφτούμε μια απόδοση επί των επενδύσεων και αυτό είναι σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι συνήθως η οικονομική βάση των επιχειρήσεων αυτών είναι αρκετά δυνατή αλλά όχι τόσο δυνατή ώστε να μπορούν να επιβιώσουν 5 έως 10 χρόνια χωρίς να έχουν απόδοση από τις δραστηριότητες τους. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε όλα μας τα χρήματα σε έρευνα και τεχνολογία. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα βελτιστοποιήσουμε την κατάσταση ούτως ώστε να έχουμε κάποια υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποια υποστήριξη σε σχέση με μεγαλύτερα προγράμματα στα οποία θα μπορούσαμε να ενταχθούμε ε, ε, σε, ε, εφόσον είμαστε οντότητες εξειδικευμένες έχουμε έναν κίνδυνο, αλλά όταν μιλήσουμε για ε, κίνδυνο ε, και κατανομή των εσόδων, ο κίνδυνος είναι, όπως είπα, ο κίνδυνος να μπούμε σε μεγάλα προγράμματα ε, και ως προς τα έσοδα θα έρθουν σε 5-10 χρόνια. Τώρα η αγορά η, στην άμυνα. Έχουμε και την αγορά την μη στρατιωτική, αλλά η αγορά η αμυντική Έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση όπου έχουμε προϋπολογισμούς που μειώνονται, έχουμε προγράμματα που έχουν φτάσει στο επίπεδο οριμότητας ή βρίσκονται λίγο πριν από το επίπεδο οριμότητας στο FAS 4 Ευρώπη το θέμα των ε, δορυφόρων που έχουμε στην Ευρώπη και δεν βλέπουμε μεγάλα προγράμματα στον ορίζοντα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο για τις μικρομεσαίες να σκεφτούν τι θα φέρει το μέλλον. Αν δεν έχουμε σήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα διάφορα εθνικά όργανα ότι θέλουν να έχουν κάποια ανάπτυξη και θέλουν να επιδιώξουν μερικά νέα προγράμματα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των τεχνολογιών περαιτέρω, τότε η κατάσταση είναι δύσκολη στον, στην άμυνα. Έχουμε ένα, μια αγορά με πολλή ρύθμιση αν είστε στην αγορά θα είστε και στην αγορά, αλλά αν θέλετε να εισέρθετε σε αυτή την αγορά έχετε να αντιμετωπίσετε ορισμένα εμπόδια και φραγμούς. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα βελτιστοποιήσουμε την πρόσβαση ε, στις διάφορες δυνατότητες αγοράς ε, που εμφανίζονται στον ορίζοντα. Όπως είπα, δεν έχουμε νέα ε, εθνικά προγράμματα λόγω των υψηλών επενδύσεων που απαιτούνται και της χαμηλής δραστηριότητας στην αγορά. Αλλά από την άλλη πλευρά αν δούμε τον τομέα των οπλισμών και τον ε, ναυτικό τομέα, ε, δεν έχουμε μερικές από τις δραστηριότητες που μπορούν να αποφέρουν και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε νέα προγράμματα που θα ε, δίνουν περισσότερη σημασία σε αυτού του είδους τις εφαρμογές. Παραδείγματος χάρη, τα κέντρα που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να συγκεντρώσουμε τους διάφορους τύπους αεροσκαφών, ελικοπτέρων ε, ε, στον, ίδιο χώρο, στον ίδιο ευρωπαϊκό, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Θα πρέπει λοιπόν να προβάλλουμε ιδέες για να εξασφαλίσουμε αυτούς τους χώρους που είναι διαθέσιμη για τα διάφορους τύπους αεροσκαφών και να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση και αν εξετάστε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές νέες εξελίξεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτές τις δραστηριότητες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έχει κάνει πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια, αλλά και μερικές δραστηριότητες υλιοποιήθηκαν ε, για την μελλοντική βοήθεια στην Ευρώπη και χαίρομαι που ήμουνα σε αυτήν την ομάδα που ε, προσανασβελιζόταν περισσότερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα μπορείτε να βρείτε μερικά επιχειρήματα για τις δυνατότητες που κινδυνεύουμε να χάσουμε και επίσης ε, για τις δυνατότητες που θα έπρεπε να ενισχύσουμε, να προωθήσουμε και αυτός ε, είναι ένας ε, τομέας ε, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις με αποδοτικό τρόπο. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα παγιώσουμε την ζήτηση στην Ευρώπη. Γιατί σκεφτόμαστε ατομικά προγράμματα, πρέπει αυτά να συγχωνευθούν για να ικανοποιήσουν ανάγκες ενός μεγαλύτερου προγράμματος και να συγκεντρώσουν όλες αυτές τις ιδέες για την ενοποίηση και παγιοποίηση της ζήτησης. Θα πρέπει να έχουμε κοινά προγράμματα και να συμφωνήσουν όλες, όλα τα εθνικά όργανα. Επίσης, κοιτάζουμε πέραν του Ατλαντικού, μιλάμε για το πολλά χρήματα που ξοδεύονται εκεί στις Ηνωμένε για την άμυνα και την ασφάλεια. Και λέμε ότι θα πρέπει να, στο ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχουν περισσότερα κονδύλια για τις δραστηριότητες. Αλλά αν συγκρίνουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε, θα δούμε ότι εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε λιγότερα χρήματα. Αλλά αν εξετάσετε τα συστήματα και τα επιτέρατά μας και την τεχνογνωσία που αναπτύξαμε, θα δείτε ότι δεν έχουμε καθυστέρηση, δεν βρισκόμαστε πίσω. Εκεί που βρισκόμαστε πίσω είναι στα μεγάλα προγράμματα. Πρέπει λοιπόν αυτό που είπα να ενοποιήσουμε και να εδραιώσουμε τη ζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίπεδο για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες που έχουμε για αυτού του είδους τα προγράμματα. Η ορθολογικοποίηση της ζήτησης είναι περίπλοκη διαδικασία, πολλές προδιαγραφές χρειάζονται, ίσως μπορεί να υπάρχει κάποια διευκόλυνση για το μέλλον. Η οικονομική υποστήριξη για τις μικρομεσαίες είναι κάτι που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η οικονομική χρηματοδυτική ε, στήριξη λένε δεν πρέπει να πηγαίνει προς τις μικρομεσές επειδή δεν έχουν κεφάλαια, δεν μπορούν να πληρώσουν από μόνες τους. Ότι εγώ νομίζω όμως ότι πρέπει η υποστήριξη αυτή να πηγαίνει προς τις μικρομεσαίες. Μίλησα για τον κίνδυνο, τα έσοδα, για τα μεγάλα προγράμματα. Αν σκεφτούμε λοιπόν τα μεγάλα προγράμματα, ε, χρειάζεται μια προκαταβολή, με χρήματα εκ των προτέρων για να προχωρήσει η βάση των μικρομεσαίων. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ορισμένα χρήματα για να αρχίσουμε ορισμένα προγράμματα και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας όταν μιλάμε για την κοινή πολιτική ασφάλειας και έρευνας για την διτή διπλή χρήση αν έχουμε όλα την προσέγγιση, την κοινή προσέγγιση επιστοποίηση, όλα αυτά σχετίζονται με τις ε, μικρομεσαίες. Ε, Θα πρέπει λοιπόν να συγχρονίσουμε τις προσπάθειές μας και να έχουμε ενοποίηση και δρέωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φτάνω έτσι στα συμπεράσματά μου. Οι δράσεις είναι απαραίτητες για την εκκίνηση προγραμμάτων βάσει ενός συντονισμένου προγράμματος για να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική προσέγγιση με ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη βιομηχανικών δυνατοτήτων. Να μην τις χάσουμε, διότι αν τις χάσουμε σήμερα δεν θα τις ανακτήσουμε πλέον, διότι θα βρεθούμε ε, σε πολύ ε, κακή ανταγωνιστική θέση σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε και την ασιατική αγορά και αν χάσουμε αυτές τις δυνατότητες δεν θα τις ανακτήσουμε διότι δεν θα μπορούμε ε, να χρηματοδοτήσουμε τις χαμένες δυνατότητες. Θα πρέπει λοιπόν να να ταινίσουμε το μέλλον με εμπιστοσύνη, θα είναι λαμπρό ε, τότε στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Θα πρέπει να έχουμε ε, μια συνεχή επένδυση σε έρευνα ε, και ανάπτυξη, διότι δεν θα υπάρξουν νέα προγράμματα. Τι θα κάνουν εντωμεταξύ οι μικρομεσαίες αν δεν υπάρχουν νέα έργα και προγράμματα. Θα πάνε προς άλλες κατευθύνσεις, θα αφήσουν ορισμένους τομείς και πάλι θα χάσουμε δυνατότητες η βελτίωση της συνεργασίας, η χρησιμοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο σε μελλοντικά προγράμματα ανάπτυξης, θα πρέπει να υπάρχει αξιοπιστή εμπιστοσύνη και τέλος θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις γεωστρατηγικές προτεραιότητες σε ένα νέο πλαίσιο. Αν δούμε λοιπόν την άμυνα στον κυβερνοχώρο είναι νομίζω ε, νέα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Θα πρέπει να δούμε πόσα θα βελτιώσουμε το περιβάλλον μας και όχι μόνο να μιλάμε γι' αυτό. Θα πρέπει να μην έχουμε ε, διαρροές προς τη λαθεσμένη κατεύθυνση. Θα πρέπει να έχουμε τη δύναμη να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Ζούμε σε μια ασφαλή κοινωνία, αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε ένα επίπεδο δραστηριοτήτων να μην υπάρχει διάβρωση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών δυνατοτήτων. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα έχουμε την βάση, την ευρωπαϊκή ε, τεχνολογική και βιομηχανική αμυντική βάση. Πρέπει να την ενισχύσουμε και να έχουμε νέους τύπους δραστηριοτήτων. Με δυνατή πολιτική βούληση πέραν των θετικών δηλώσεων, δηλαδή για συγκεκριμένα ε, αποτελέσματα, πρέπει να προχωρήσουμε διότι αυτό θα είναι υπέρ της σταθερότητας της βιομηχανίας μας. Θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης και τον ε, κώδικα ε, δεοντολογίας που θα έχουμε. Αν είμαστε στον τομέα της άμυνας, πολλοί λένε ότι δεν είμαστε ηθικοί, διότι δεν είναι ηθική η άμυνα και θέλω να σας ρωτήσω εάν ε, ε, με την ε, τρομοκρατία ε, που έχουμε απέναντί μας, αν βλούμε τι συμβαίνει στον κόσμο μας όπου θέλουμε να συνεργαστούμε με τις χώρες για να τις καθησυχάσουμε, τότε είναι απαραίτητο στο μέλλον να ασχοληθούμε με τον τομέα της ασφάλειας και άμυνας και να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες μας προς την κατεύθυνση αυτή και να σκεφτούμε την δεοντολογία στον τομέα μας που ενδιαφέρει πολύ τους πελάτες μας ε, στην όλη αλυσίδα. Έχουμε ομάδα δεοντολογίας και σκεφτόμαστε ποια είναι η δεοντολογία και πόσο μπορούμε ε, να γίνουμε επιχειρήσει ε, κατάλληλες στα νέα προγράμματα και προσπαθούμε να εντάξουμε αυτές τις ηθικές απόψεις. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι έχουμε δώσει τόση σημασία στις μικρομεσαίες στα τελευταία 20 χρόνια ούτως ώστε ε, να ακολουθήσουμε ε, ό,τι γίνεται στον τομέα ασφάλειας και άμυνας. Νομίζω ότι έχουμε καλό επίπεδο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νομίζουμε ότι αξίζει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση με ηθική βάση, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα αιτήματα των διαφόρων εθνικοτήτων, να τα ενοποιήσουμε, να ενοποιήσουμε τη ζήτηση και θα, με χαρά θα ε, σας συνεργαστούμε μαζί σας ως οργάνωση ASD, διότι νομίζουμε ότι αξίζει. Ακούσαμε την ε, αρμόδια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Άμυνας το πρωί τώρα θα ακούσουμε τον ομόλογό της από την ίδια βέβαια υπηρεσία το απόγευμα, τον κύριο Γκος. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας για να συζητήσω τις δυνατότητες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Και θα ήθελα να δούμε και πέρα από το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό για τα θέματα της άμυνας. Κάποια από τα πράγματα που θέλω να πω θα επαναλάβουν ουσιαστικά αυτά τα οποία είπε ο κ. Σάλερς, αλλά η επανάληψη μερικές φορές είναι χρήσιμη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο σκελετός, θα έλεγα, της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης. Έχουμε στην Ευρώπη, στον τομέα των πολιτικό και στρατιωτικό, 20 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 97% των, των, της βιομηχανικής παραγωγής τα δύο τρίτα συνολικά των θέσεων απασχόλησης. Οι αριθμοί είναι τεράστιοι. Αντιπροσωπεύουν το 58% της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Υπάρχουν επιχειρήματα λοιπόν για ισχυρές, αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές ε, μικρομεσαίες βιομηχανίες. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες καινοτομίας και έρευνας. Ήδη από το 2007 το είπαν οι Υπουργοί Άμυνας η μελλοντική τους επιτυχία λοιπόν θα εξαρτηθεί από την σωστή χρήση αυτών των δυνατοτήτων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτό θα γίνει λοιπόν, μπορεί να γίνει στην Ευρώπη και μπορεί να γίνει στις μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι σχέσεις, ε, μάλλον οι επιχειρήσεις οι οποίες στρέφονται στον τομέα της άμυνας ε, ε, βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη, βέβαια υπάρχουν σε κάποιες περιφέρειες κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Ε, ε, υπήρξαν αναφορές και στην παρουσίαση της κυρίας Άστον και στην παρουσίαση της Επιτροπής αργότερα, αλλά αυτά θα τα πει ο επόμενος ομιλητής. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάρα πολύ συχνά αντιμετωπίζουν και εμπόδια έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται τις επιχειρηματικές ευκαιρίες της ευρωπαϊκής αγοράς διαθεσιμότητα πληροφόρησης, γραφειοκρατικά εμπόδια, βελτίωση της εικόνας τους. Βασικά πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να τις γνωρίζουν. Αυτά λοιπόν έχουν ήδη αναγνωριστεί και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την ανακοίνωση για τις μικρές λεγόμενες επιχειρήσεις, η οποία όμως ανακοίνωση δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες για την άμυνα. Εδώ έχουμε μια διαφορετική διάσταση, μια επιπλέον διάσταση. Έχουμε βέβαια μια γενική διεύθυνση η οποία ασχολείται με αυτά τα θέματα. Αυτή η επιπλέον διάσταση ε, θα πρέπει να δίνει περισσότερες ευκαιρίες ε, στις μικρομεσαίες. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο και θα επανέλθω. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν σαν ευρωπαϊκή βιομηχανία, ε, σαν υπηρεσία μάλλον στον τομέα αυτό. Εμείς προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη που είναι οι άνθρωποι που μας ελέγχουν με τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες για να βελτιώσουμε τη θέση τους στον τομέα τον αμυντικό. Αυτό δεν είναι καινούριο. Ήδη από το 2009 είχαμε δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη των μικρομεσαίων στην αμυντική βιομηχανία αντιμετωπίζοντας τα θέματα των ίσων ευκαιριών για τις υπεργολαβίες ελάχιστος χρόνος αντίδρασης, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, ενίσχυση της βιομηχανικής συνεργασίας, κοινωνικές διαστάσεις και ε, νέες τεχνολογίες. Απαιτείται όμως να ενταθούν οι προσπάθειες και γι' αυτό το πρόγραμμα δράσης για τις μικρομεσαίες έγινε δεκτό και από τους Γενικούς Γραμματείς των Αρμόδιων Υπουργείων τον μήνα Μάρτιο. Θα υποστηριχθούν λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βελτιώνοντας ε, την ε, κυκλοφορία της πληροφορίας, ε, ενισχύοντας την καινοτομία, διευκολύνοντας την, τις ρυθμίσεις, τις διακανονιστικές στον τομέα των εργολαβιών κτλ. Να αναφερθώ σε κάποιες πιο συγκεκριμένες δράσεις. Καταρχάς, ε, ενημέρωση για τις επιχειρηματικές δυνατότητες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν το δυναμικό, το προσωπικό και τα χρήματα να ελέγχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλους, όλες τις ευκαιρίες τις επιχειρηματικές. Γι' αυτό λοιπόν εμείς στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας ξεκινήσαμε ένα πόρταλ στον ιστότοπό μας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Με λίγα κλικ μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να γνωρίσει όλες τις επιχειρηματικές βιομηχανίες σε σχέση με τις προμήθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Ένα one-stop shop. Τώρα για την έρευνα και την ανάπτυξη οργανώνονται πάρα πολλές συναντήσεις ανάμεσα στις βιομηχανίες, φέρνουμε σε επαφές τις βιομηχανίες σε διαμεθοριακό επίπεδο ε, να προχωρήσουν σε κοινά επενδυτικά προγράμματα. Προγράμματα όπου όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεισφέρουν. Δεύτερον, διευκολύνουμε ή προσπαθούμε να διευκολύνουμε και την πρόσβαση στα κοινοτικά χρήματα. Ε, ίσως πολλές φορές είναι περίπλοκο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Απαιτείται να γνωρίζουν το θεσμικό περιβάλλον, να καταθέτουν σωστές αιτήσει και ακριβώς εμείς προσπαθούμε να διευκολύνουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποστηριχθούν μέσα από ομάδες εργασίας στα διάφορα κράτη-μέλη ή τοπικές βιομηχανίες. Φέτος οργανώσαμε τέτοιες συναντήσεις στην Αυστρία και του χρόνου αν κατάλαβα καλά θα υπάρξει ε, μια συνάντηση στην Πολωνία για τις χώρες του Βίσεγκραντ και αν πράγματι οι βιομηχανίες δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με μας, μπορούμε εμείς να πάμε σε αυτούς και να τους εξηγήσουμε σε αιτήσια βάση το τι συμβαίνει. Ενισχύουμε και πιλωτικά προγράμματα που προσελκύουν διαφορετικά ταμεία στην Πολωνία, στην Πορτογαλία. Υπάρχουν δύο πολύ πετυχημένα προγράμματα που είναι το πρώτο βήμα για τον καθορισμό μιας πιο συστηματικής στήριξης η οποία θα παρέχει ε, βοήθεια σε τακτική βάση και θα επιτρέπεται έτσι στις επιχειρήσεις αυτές τις χώρες να χρησιμοποιούν τα χρήματα των περιφερειακών ταμείων. Πρέπει εδώ να τονίσω το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα υπάρχοντα μέσα και με τα μελλοντικά μέσα για την ευημερία θα έλεγα των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα για την ανταγωνιστικότητα, για την συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις κτλ. Και να διασφαλίσουμε επίσης και τη συμπληρωματικότητα με τον ΝΑΤΟ. Δεν πρέπει να κάνουμε επικαλύψεις. Γιατί έχουμε λίγα χρήματα για να το κάνουμε. Είναι ξεκάθαρη η βούληση των κρατών μελών έτσι ώστε οι συνέργειες αυτές από να γίνουν ουσιαστικές. Η υποστήριξη στις μικρομεσαίες θα πρέπει να είναι έγκαιρη και εύθετη, όπως είπε και ο κύριος Άλευς, και γι' αυτό αναπτύξαμε ακριβώς ε, ένα κατάλογο κρίσιμων τεχνολογιών ε, στα διάφορα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μην είμαστε εξαρτημένοι στο μέλλον από στρατηγικής φύσεως ε, βιομηχανίες εκτός Ευρώπης. Υπάρχουν τομείς τους οποίους θα πρέπει να προχωρήσουμε στην Ευρώπη, το ΣΕΖΑΡ σαν παράδειγμα, τηλεκατευθυνόμενα μέσα και υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες με συγκεκριμένους τρόπους, σε συγκεκριμένους θύλακες θα έλεγα, μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ικανότητες που υπάρχουν. Υπάρχουν επίσης και προτεραιότητες στην απόφαση για χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Αυτό είναι ένα πρώτο, ένας πρώτος τομέας αν θέλετε. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μας το πει αργότερα είναι να δώσει μια σωστή ευκαιρία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και όχι απλά ένα συγκεκριμένο κομμάτι της πίτας από την διαθέσιμη χρηματοδότηση. Πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις αγορά διαμεθοριακά και σε διεθνές επίσης επίπεδο, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό. Εμείς σαν Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία είναι να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε με άμεσο τρόπο τις μικρομεσαίες, να τις ενημερώσουμε σωστά ε, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια. Ευχαριστώ κύριε Γκούς και για τα καλά σας λόγια για την δική μου χώρα, την Πολωνία και για τα προγράμματα που εξελίσσονται στη χώρα μου. Ο κ. Τοκάρσκι, Πολωνός συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως ακούσαμε από τους δύο προηγούμενους ομιλητές είναι καθοριστικός στον αμυντικό τομέα. Εγώ θα περιοριστώ σε θέματα που αφορούν τη δική μας διεύθυνση, καθώς και τις δράσεις τις οποίες θέλουμε να αναπτύξουμε για να στηρίξουμε το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον αμυντικό τομέα. Βεβαίως αυτά που έχω να σας πω συμβαδίζουν κατά πολύ με αυτά που ήδη ακούσαμε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά όχι μόνο, πλήττονται από τον κατακαιρματισμό της αγοράς, έχουν δύσκολη πρόσβαση στις αγορές των άλλων χωρών και των τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι σήμερα ακόμα πιο οξύ σαν πρόβλημα, καθότι βλέπουμε περικοπές στον αμυντικό προϋπολογισμό όλων των χωρών και αυτό δείχνει πόσο ευάλωτες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μια, σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον η πρόσβαση στην αγορά, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες. Ο κατακαιρματισμός της αγοράς είναι βεβαίως προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς. Είναι κάτι που ίσως ενισχύει ακόμη πιο πολύ αυτό που ακούσαμε, που είναι κάτι που αφορά την δεοντολογία καθώς και την ε, εικόνα στην κοινή γνώμη αυτών των επιχειρήσεων. Πολλές ε, φορές βλέπουμε ότι στον τομέα αυτό το θέμα της δεοντολογίας είναι κάτι που προβληματίζει πολύ την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Τώρα, ποια είναι τα θετικά αυτού του τομέα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι μικρομεσαίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας βρίσκονται σε μία πολύ, ε, αν θέλετε, καινοτόμα βιομηχανία βρίσκονται σε, στην πρωτοπορία της τεχνολογίας. Αυτό είναι το θετικό, πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Πολύ καινοτομία και καινοτόμες σκέψεις, νέες τεχνολογίες προκύπτουν από αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δίνουν δυνατότητες ανάπτυξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον αμυντικό τομέα. Τι προτείνουμε λοιπόν εμείς. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αμυντικό τομέα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τις δυνατότητες που παρέχονται στις ε, επιχειρήσεις αυτές που δραστηριοποιούνται στον μη αμυντικό τομέα. υπάρχει σήμερα γνώση αυτών των εργαλείων, αυτών των δυνατοτήτων και εξετάζουμε τις δυνατότητες να επεκταθεί αυτή η χρήση και σε επιχειρήσεις που ε, ενεργοποιούνται είτε αποκλειστικά και μόνο στον ε, στρατιωτικό τομέα, είτε είναι παρούσες και στην ε, πολιτική αεροπορία ή δραστηριοποιούνται και στον μη στρατιωτικό τομέα με μία προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τους θύλακες, την κατακαιρματισμένη αγορά που χαρακτηρίζει τον αμυντικό τομέα, τον τομέα των εξοπλισμών. Επίσης θα θέλαμε να βοηθήσουμε αυτή την στρατηγική των συνεργατικών σχηματισμών, των θυλάκων μέσα σε μεγαλύτερους θύλακες και θα προσφέρουμε ένα νέο εργαλείο για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 2014. Οι πρώτες δυνατότητες χρηματοδότησης θα είναι διαθέσιμες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2014, την Άνοιξη και βεβαίως θα συνεργαστούμε με τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Άμυνας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλουν ε, αιτήσει και να συμμετάσχουν στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση. Η τελευταία τέτοια δυνατότητα χρηματοδότησης ήταν πολύ επιτυχής. Δεν έχω ακριβή στοιχεία, αλλά ε, η χρηματοδότηση ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δύο, πρέπει να σας πω, τέτοιες προσπάθειες χρηματοδότησης ήταν επιτυχής. Θέλουμε λοιπόν να επεκτείνουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης και στους ε, εμπλεκόμενους στον τομέα των εξοπλισμών, τον αμυντικό τομέα. Επαναλαμβάνω, αυτοί οι συνεργατικοί σχηματισμοί θα πρέπει να υποφεληθούν. Έχουμε σήμερα επίσης και ένα νέο συντονισμό για την επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όλα αυτά προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αμυντικού τομέα στην Ευρώπη. Τρίτον, ο κύριος Γκος μίλησε για την καλύτερη πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία, στην χρηματοδότηση μέσω διαρθρωτικών ταμείων. Και αυτό προσπαθούμε να το διευθετήσουμε με δύο τρόπους και βεβαίως αυτό το κάνουμε συνεργαζόμενοι με τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία, βελτιώνοντας ε, τα δίκτυα, τις έξυπνες στρατηγικές, όχι μόνο για να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, αλλά αυτή η στρατηγική έχει σαν σκοπό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να οδηγήσει για τα επόμενα 7 χρόνια σε καλύτερη χρηματοδότηση μέσω των περιφερειακών ταμείων. και αυτό προσπαθούμε να το ενσωματώσουμε σε αυτήν την έξυπνη ε, στρατηγική. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια σειρά συναντήσεων με δέκα διαφορετικές περιφέρειες, οι οποίες έχουν δείξει ενδιαφέρον. Κάποιες μάλιστα έχουν προετοιμάσει προτάσεις για την ε, χρήση όλων αυτών των δυνατοτήτων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο στον ε, ε, στρατιωτικό βιομηχανικό τομέα, αλλά και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και εκτός της αμυντικής βιομηχανίας. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τους καλύτερους τρόπους έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες στον στρατιωτικό και μη στρατιωτικό τομέα. Βεβαίω, καταρχήν πρέπει να αποσαφηνηθούν οι κανόνε. Σήμερα υπάρχουν ε, μικρομεσαίες επιχειρήσει οι οποίε είτε διστάζουν να υποβάλουν αιτήσει για χρηματοδότηση, είτε οι αιτήσει του δεν προχωρούν. Οι κανόνες πολλές φορές δεν είναι σαφείς και θέλουμε να τους αποσαφηνίσουμε, θέλουμε να δημοσιεύσουμε ένα εγχειρίδιο που με πολύ σαφή τρόπο παρουσιάζει αυτές τις προϋποθέσεις, πώς μπορεί ένα πρόγραμμα να χρηματοδοτηθεί. Ο κύριος Γκος ανέφερε αυτή τη δυνατότητα. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πιλωτικές προσπάθειες οι οποίες στηρίζονται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας έτσι ώστε να γενικευθούν. Τέλος, και σε σχέση με αυτά που ήδη ακούσαμε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε άλλους τομείς. Υπάρχει το πρόγραμμα μέχρι το 2020, εκ των οποίων η χρηματοδότηση, το, 20% συγγνώμη, της χρηματοδότησης απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τις ε, επιχειρήσεις αυτές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον αμυντικό τομέα υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω πρόσβασης στην χρηματοδότηση γιατί έχουμε αναλύσει τις δυνατότητες ανάπτυξής τους για τα επόμενα 10-20 χρόνια και είναι πολύ ενθαρρυντικές στον τομέα της ε, πολιτικής ε, αεροπορίας, παραδείγματος χάριν, όπου ο εξοπλισμός για την αύξηση της ασφάλειας των πτήσεων είναι κάτι που δίνει νέες δυνατότητες ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα αυτό και βεβαίως η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Βεβαίως σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τη δράση μας, να βελτιστοποιήσουμε τις προσπάθειές μας και βεβαίως πιστεύουμε ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου θα οδεύουν προς αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Ο κύριος Γκάλερ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι εισηγητής για την έκθεση βάσης εξοπλισμών στην Ευρώπη και βεβαίως ε, εδώ υπάρχει η ημερομηνία του Δεκεμβρίου και της συνάντησης κορυφής. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντική η ακρόαση που διοργανώσαμε σήμερα καθότι μας χρειάζεται σήμερα ένα πλαίσιο και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε η βιομηχανική βάση της Ευρώπης να ενισχυθεί και οι δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν και να αναπτυχθούν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βεβαίως ε, είναι για μας ε, καθοριστικές. Θέλουμε να τις στηρίξουμε. Ξέρουμε τι δυνατότητες στην απασχόληση υπάρχουν από την στήριξη των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά βεβαίως όπως ξέρετε ο τομέας ε, ο αμυντικός ε, έχει λίγους πελάτες. Οι πελάτες είναι κυρίως τα κράτη, οι εθνικές αρχές. Βεβαίως υπάρχουν προϊόντα, εξοπλισμοί, τεχνικοί εξοπλισμοί που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από τον μη στρατιωτικό τομέα, όπως η επικοινωνία, τα ηλεκτρονικά συστήματα, ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από τις δυνάμεις ασφαλείας εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά βεβαίως αυτό που μας απασχολεί εδώ είναι όταν ε, η βάση των πελατών, αν θέλετε, είναι τόσο περιορισμένη, όταν ο βασικός πελάτης αυτή, αυτού του τομέα είναι το κράτος, είναι πολλές φορές δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τις στρατιωτικές από τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό βλέπετε δυνατότητες να δείτε μία αν θέλετε ελάφρυνση των διαδικασιών και περισσότερη ευελιξία. Ξέρουμε σήμερα, παραδείγματο χάρη, ότι αυτές οι πολύ ευαίσθητες τεχνολογίες πολλές φορές προστατεύονται σε υπερβολικό βαθμό. Πώς μπορεί το κράτος, αν θέλετε, το οποίο είναι αυτός ο οποίος δίνει την εντολή, παραγγέλνει έναν εξοπλισμό, να δείξει ότι είναι διατεθειμένο να μοιραστεί αυτή τη τεχνολογία με άλλους τομείς και πώς είναι δυνατόν να εξορθολογικοποιήσουμε λιγάκι τις απαιτήσεις, τη ζήτηση έτσι ώστε να διοχετευθούν τα προϊόντα αυτά και σε άλλους τομείς όταν ο εντολοδόχος αν θέλετε είναι το κράτος, πολλές φορές ξέρουμε πόσο άκαμπτη είναι η διαδικασία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που ξέρετε, σύμφωνα με την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι ο τομέας αυτός μπορεί να βρει νέες δυνατότητες ανάπτυξης Εάν λίγο εξισορροπηθεί η προσφορά και η ζήτηση, ξέρουμε σήμερα ότι οι τιμές παραδείγματος χάρη ανάπτυξης αυτών των προγραμμάτων είναι εξαιρετικά υψηλές και αυτό είναι και κάτι το οποίο καθορίζεται από την σχέση που έχουμε σήμερα προσφοράς και ζήτησης. Υπάρχει δυνατότητα λίγο να μαλακώσει αυτό το σύστημα, να υπάρξει περισσότερη ευελιξία βάσει της εμπειρίας σας. Μπορείτε να μου πείτε όχι. Υπάρχουν συμφωνίες, εμείς έχουμε συγκεκριμένες προθεσμίες για την ε, ε ολοκλήρωση μιας διαδικασίας παραγωγής, συγκεκριμένες τιμές και δεν πρόκειται να παρεκκλίνουμε καθόλου από αυτό. Είτε μπορείτε εσείς να διαπιστώσετε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το α400 μη σήμερα έχει φτάσει μία τιμή τόσο υψηλή σε σύγκριση με άλλα παρόμοια προϊόντα που ε, θα πρέπει κάπως να δικαιολογηθεί και να στηριχθεί. Και σας έδωσα ένα μόνο παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης. Αυτά προς το παρόν. Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά ίσως ε, θα περιμένω για να τις κάνω λίγο αργότερα. Ευχαριστώ πολύ, Μάικλ. Η κυρία Κοπά. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ευχαριστώ για αυτήν τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε τι μπορούμε να περιμένουμε από τη Σύνοδο Κορυφής εμείς ως Κοινοβούλιο. Εσείς τι περιμένετε ως συγκεκριμένα αποτελέσματα από το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Διότι ξέρουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής ήταν αρκετά φιλόδοξη ε, και υπάρχει από πλευράς ε, των ε, πρωτευουσών επιφύλαξη. Τι περιμένετε, τι φοβάστε κατά κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Γερέκης. Ευχαριστώ πολύ. Ένα πράγμα είναι προφανές. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό ε, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως για να μπορέσουν να συνεργαστούν με δομές ε, διεθνικές. Στο παρελθόν βρισκόμασταν σε μια κατάσταση όπου υπήρχαν μεγάλοι όμιλοι και αυτοί οι μεγάλοι όμιλοι είχαν τα πάντα, είχαν τα όσα χρειαζόντουσαν. Μετά ε, παρήγαν διάφορα αγαθά, ό,τι ήταν αναγκαίο για να ε, όλα τα προϊόντα που χρειαζόντουσαν στον τομέα της άμυνας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και συνεπώς τώρα υπάρχει αυτό το outsourcing, αυτή η ανάθεση προς τα έξω, η υπεργολαβία με έναν μεγάλο αριθμό υπεργολάβων αλλά νομίζω ότι υπάρχει εδώ μια σύγκρουση ανάμεσα στις δομές. Υπάρχουν οι μεγάλες δομές, οι οποίες είναι κλειστές, που συχνά είναι εθνικές ή πολυεθνικές και από την άλλη πλευρά υπάρχουν ε, οι μικρές επιχειρήσεις αδύναμες από οικονομικής πλευράς, αδύναμες ως προς την ικανότητα να προστατεύσουν ε, την πνευματική τους ιδιοκτησία. Πρέπει να βρεθεί νομίζω μια λύση σε αυτό το πρόβλημα μια λύση που θα επιτρέψει την εξασφάλιση μιας νομικής ασφάλειας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα επιτρέψει την εξασφάλιση κάποιας χρηματοδότησης των μικρομεσαίων σε αυτόν τον τομέα και επίσης θα επιτρέψει την προστασία των κρατών. Και αυτό που θέλουν να κάνουν ε, ε, μυστικά, διφόσον πολύ συχνά τα θέματα αυτά είναι απόρριτα, είναι μυστικά και υπάρχει και το θέμα του συντονισμού που τίθεται. Κατά τη γνώμη μου, ένα νέο κείμενο νομικό, νέοι κανόνες για τις ε, μικρομεσαίες θα ήσαν αναγκαίες για να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας, είναι μόνο ε, χρηματοοικονομικές, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία και άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλει, κανείς να, θέλει να συμπληρώσει ο κύριος Γκαλέρ. Ναι όσον αφορά την συζήτηση για την πιστοποίηση καθώς ε, και το χρόνο που έχει άμεση σχέση με τον καθορισμό της τιμής. Εσείς, σαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων που παράγει, υπάρχει ένας πραγματικός, ρεαλιστικός παράγοντας χρόνου και τιμής. Μπορείτε να τον καθορίσετε κάπως, να τον ορίσετε. Όσον αφορά την πιστοποίηση, κανονικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να, ισχύει η ίδια, να ισχύουν οι ίδιες Η πιστοποίηση λοιπόν θα είναι κάτι το απλό από ό,τι καταλαβαίνω. Πρόεδρος, σας δίνω λίγα λεπτά, maximum πέντε, για να απαντήσετε. Μπορείτε να απαντήσετε σε όποια ερώτηση θέλετε και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τοκάρσκι. Ευχαριστώ. Διορθώστε με κύριε Γκάλερ. Η ερώτησή σας έλεγε ότι αν υπάρχει κάτι στην άποψη που έχουν ε, τα κράτη-μέλη σχετικά με τις δαπάνες που θα μπορούσε να αλλάξει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας πολύ συχνά αναζητούμε εναλλακτικούς τρόπους για προγράμματα τα οποία όταν είναι ας πούμε συνεργατικά, όταν είναι προγράμματα που εμπλέκουν πολλούς εταίρους, μερικές φορές έχουν υψηλό κόστος. Η, εμπειρία σαν παράδειγμα του μεταγωγικού αεροσκάφους Α400 μη δεν ήταν αρνητική. Συνεργαστήκαμε φυσικά και με τις ιδιωτικές εταιρείες, με το ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο επιτάχυνε γενικά τις διαδικασίες πιστοποίησης του αεροσκάφους και έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για θετικά στοιχεία ακριβώς λόγω της συνεργατικής φύσης της εξέλιξης του αεροσκάφους. Η αναζήτηση νέων τέτοιων σχεδίων και η τοποθέτησή τους σε ένα υγιές πλαίσιο εξ αρχής, γιατί γνωρίζουμε ότι σε προγράμματα αντίστοιχα συνεργατικά στο παρελθόν η κατάσταση άλλαξε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του αεροσκάφους και αυτό οδήγησε σε καθυστερήσεις, σε υπερβολικό κόστος κτλ. Υπάρχουν κάποια προγράμματα τεχνικά καινοτόμα στα οποία δεν υπάρχει ιδιαίτερος ανταγωνισμός και εκεί μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να εναρμονίσει σε επίπεδο κρατών μελών πάντα τις τεχνικές απαιτήσεις και τις τεχνολογικές δυνατότητες έτσι ώστε με μειωμένο σχετικά κόστος να υπάρξει προστιθέμενη αξία για την παραγωγή των απαιτούμενων μέσων. Για την κυρία Κοπά και τι περιμένουμε από το Συμβούλιο. Από πλευράς μας, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομίζω ότι θέλουμε να προχωρήσουν στον τομέα της standardization, της πιστοποίησης, των μικρομεσαίων, της διτής χρήσης, της έρευνας και τέλος να τεθεί ε, υποσυζήτηση το θέμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ε, είναι ένα τομέα στον οποίο μπορεί να υπάρξει περαιτέρω συνέργεια. Και τέλος να απαντήσω στην τελευταία ερώτηση, πολύ συχνά στις συζητήσεις που έχουμε με τα κράτη-μέλη, διακρίνουμε ένα φόβο. Αν πράγματι υπάρχει δηλαδή μια σωστή ολοκλήρωση ε, στον τομέα της αγοράς και χρειάζεται να κλείσουν μονάδες και τα λοιπά. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα κερδίσουν και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα χάσουν. Ε, τα κράτη-μέλη δηλαδή έχουν ένα φόβο ε, προς την κατεύθυνση αυτή αν υπάρξουν περαιτέρω ε, ολοκληρώσεις στην βιομηχανική παραγωγική βάση, αν υπάρξουν συγχωνεύσεις κτλ. Το θέμα είναι ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό θα σημαίνει ότι κάποια τμήματα της βιομηχανίας, της αμυντικής στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα είναι οικονομικά ανταγωνιστικά. Δεν μπορεί κανείς έτσι κι αλλιώς να διατηρήσει μη ανταγωνιστικές παραγωγικές μονάδες έστω και σε εθνικό αυστηρά επίπεδο. Η ευρωπαϊκή συνεργασία με διαφορετικά πρότυπα, με διαφορετικούς τρόπους μπορεί να προσφέρει, είδαμε ότι σε ορισμένες χώρες υπάρχουν ορισμένες εξειδικεύσεις, από ολοκληρωμένα συστήματα είδαμε ότι ορισμένες βιομηχανίες έχουν αρχίσει και εξειδικεύονται στα λεγόμενα υποσυστήματα και υπάρχει γενικά προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Γκος, για τις ερωτήσεις του κύριου Γκάλα. Να πω ότι Νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή να συνεργαστούμε ανάμεσά μας. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε τέτοια παρακμή σε εισαγωγικά των προϋπολογισμών για την άμυνα. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε έτσι ώστε αυτά τα λίγα που έχουμε να μπορέσουμε να τα μοιραστούμε σωστά και να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες από ό,τι αν ήταν ο καθένας μόνος του. Από την άλλη, μπορεί να χάσει κανείς τις ικανότητες τις οποίες έχει με τις εξελίξεις και έτσι διακινδυνεύει το να χάσει επίσης ένα ουσιαστικό τμήμα της κυριαρχίας και της ελευθερίας δράσης. Η ελευθερία δράσης αναφέρεται όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου λοιπόν ο χρόνος για συνεργασία είναι τώρα. Αναφερθήκατε στο Α400M. Όταν ξεκίνησα πριν 20 χρόνια, ε, συζητούσαμε την εναρμόνιση των απαιτήσεων κάθε χώρας και το 1993 το πρώτο πρόγραμμα το οποίο προχωρήσαμε ήταν το Α400M και πέταξε επιτέλους 20 χρόνια μετά. Χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος για να προχωρήσει. Θα μπορούσε να είναι ε, πιο μικρός ο χρόνος, ναι. Θα μπορούσε να είναι φθηνότερο το μεταγωγικό αεροσκάφος, ναι. Αυτό έχει σχέση με πολιτικά θέματα, με οικονομικά θέματα, με εργασιακά θέματα, με θέματα κυριαρχίας και ελέγχου τεχνολογιών. Σιγά σιγά προχωράμε πάντως. Απαιτείται περαιτέρω συνεργασία και εφόσον συνεργαστούμε θα πρέπει να εναρμονίσουμε τις απαιτήσει μας τις επιχειρησιακές. Αν δείτε ένα άλλο πρόγραμμα, το NH90, το ελικόπτερο NH90. Υπάρχουν 20 διαφορετικοί τύποι αυτού του ελικοπτέρου. Η κατάσταση είναι δυσδιαχείριστη πλέον. Δεν μπορέσαμε να εναρμονίσουμε τις απαιτήσεις μας και αυτό παρουσιάζει ένα υψηλότατο κόστος για όλες τις χώρες μέλη. Όχι μόνο σε επίπεδο μονάδας, κόστος μονάδας αγοράς, αλλά σε επίπεδο προετοιμασίας, υποδοχής, ενσωμάτωσης κτλ. στις ένοπλες δυνάμεις. Τώρα τι περιμένει κανείς από τη συνάντηση κορυφής. Εγώ ελπίζω ότι στις συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε από πλευράς μας σαν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, κάποιες από αυτές θα μπορέσουν να γίνουν δεκτές από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Και θα θελήσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να επανέλθουν σε δύο χρόνια στα θέματα αυτά. Να μην περιμένουμε δηλαδή 6-7 χρόνια έτσι ώστε να ξαναέρθει στην ημερήσια διάταξη το θέμα της άμυνας. Η ασφάλεια και η άμυνα πρέπει να είναι στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Κορυφής σε ετήσια βάση θα έλεγα. Τώρα οι διαφορές ανάμεσα στις μεγάλες εθνικές επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάποιες διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των. Πριν ασχοληθώ με αυτό που ασχολούμαι, είχα δραστηριοποιηθεί στον τομέα της βιομηχανίας σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλεγα τότε ότι δεν με ενοχλεί τα μεγάλα προγράμματα να πηγαίνουν στις μεγάλες χώρες και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί είναι οι μόνες οι βιομηχανίες αυτές που θα τα καταφέρουν. Αν αποφασίσουν βέβαια να το κάνουν το καθένα μόνοι τους θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν. Αλλά αν αποφασίσουν όμως να λειτουργήσουν με εργολαβίες, να λειτουργήσουν με outsourcing, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξουν δυνατότητες και πρέπει να ρυθμιστεί η σχέση αυτή, όχι σε επίπεδο ε, ίσου τμήματος, ποσοστού της πίτας της διαθέσιμης κάθε φορά, αλλά σε επίπεδο ανταγωνιστικό ίσων ευκαιριών γιατί αν πράγματι ε, δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν τις ίσες ευκαιρίες ε, με όλες τις επιχειρήσεις και να πάρουν μέρος στους τεχνικούς και ε, οικονομικούς διαγωνισμούς, τότε δεν έχουν καμία τύχη στην βιομηχανία την αμυντική. Δίκαιες ευκαιρίες λοιπόν για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής Ο κύριος Άλλης, ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω γερμανικά την γερμανική ερώτηση και θα σας πω ότι καταρχήν αυτό που είπατε κύριε Γάλλαρη είναι το θέμα τι περιμένει μία επιχείρηση από το κράτος. Και βεβαίως εδώ υπάρχουν κάποια προκαθορισμένα στοιχεία, κάποιες διαδικασίες. Μιλήσατε για πειθαρχία. Ναι, τι σημαίνει πειθαρχία. Προχωρούμε πειθαρχικά, τηρούμε τις προθεσμίες, είμαστε αξιόπιστοι και λειτουργούμε με έναν αναπτυξιακό αλλά βιώσιμο αναπτυξιακό ε, τρόπο. Και το βιώσιμο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια μικρομεσαία επιχειρήση, γιατί είναι σημαντικό να μπορεί κάποιος να βασιστεί σε μια κατάσταση, να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα διακοπεί, αλλά η επένδυση που έχει γίνει σε τεχνογνωσία και τα λοιπά σε κατάρτιση να συνεχιστεί. Τώρα, αν Βεβαίως τα προγράμματα αυτά διακόπτονται αν δεν αντικαθιστώνται από νέα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να περιμένουν. Είναι επίγον να τροποποιηθούν, να προσαρμοστούν στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Είμαστε υποχρεωμένοι για να επιβιώσουμε, να προσαρμοστούμε στην ανάγκη της αγοράς. Γι' αυτό και Προσπαθούμε να στοχεύσουμε τους τομείς αυτούς που έχουν ανάγκες. Παραδείγματος χάρη, ο μηχανικός, ηλεκτρονικός τομέας. Και καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα προγράμματα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δώσουν δυνατότητες, είναι δηλαδή πολύ δύσκολη η πρόσβασή τους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ παραδείγματο χάρη με τη δική μου εταιρεία, όταν εργάζομαι στο στρατιωτικό τομέα και δεν υπάρχουν πλέον δυνατότητες, τι κάνω, στρέφομαι προς τον μη στρατιωτικό τομέα, αν όμως δω ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες που διαφαίνονται, προσπαθώ πάλι να προσαρμοστώ αλλά βεβαίως αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να χάσω τους πελάτες μου, πρέπει να υπάρξει προσαρμογή και όσον αφορά την κατάρτιση των συνεργατών μας. Καταλαβαίνετε ότι ένας συνεργάτης ο οποίος πλέον δεν έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του μπορώ να τον χάσω, να φύγει από μένα και να πάει σε άλλη εταιρεία κτλ. Τώρα, η ερώτησή σας όσον αφορά την πιστοποίηση. Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες καθότι στην Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αγγλία οι ε, διαφορετικές προδιαγραφές μας οδηγούν σε διαφορετικές ανάγκες για πιστοποίηση. Αυτό που έχει σημασία είναι όλα αυτά να εναρμονιστούν και να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε στην ανάπτυξη προϊόντων που κατά κάποιο τρόπο θα περνούν τα σύνορα ε, τα ευρωπαϊκά χωρίς πρόβλημα και να μπορούμε να συγκεντρωθούμε στις απαιτήσεις και τις ανάγκες ε, της Ευρώπης. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, το πιο βασικό είναι ότι όταν πλέον δεν υπάρχουν προγράμματα στον τομέα της άμυνας, είμαστε υποχρεωμένοι για να μην πεθάνουμε να στραφούμε σε άλλους τομείς. Κυρία ε, Κόπα, είπατε μας ρωτήσατε μάλλον τι περιμένουμε και πώς νιώθουμε την κατάσταση. Εμείς σαν τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περιμένουμε η Ευρώπη να μας δώσει συγκεκριμένες ενδείξεις για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθηθεί. Και ακούσαμε πολύ προσεκτικά ότι υπάρχουν σήμερα εργαλεία, υπάρχει χρήση δυνατοτήτων και εργαλείων, tool use στα αγγλικά, όπως μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το πιο σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι όταν υπάρχει η ανάπτυξη ενός προϊόντος για τον στρατιωτικό τομέα, να μπορεί αυτό σε κάποιες από τις ε, εφαρμογές του να χρησιμοποιηθεί και αλλού. Το tool use δηλαδή, να ξέρουμε ότι έχει συγκεκριμένες εφαρμογές στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και στον τομέα ο οποίος δεν ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους εξοπλισμούς. Θέλουμε λοιπόν να μας δώσετε ενδείξεις να μπορέσουμε οι μεγάλοι όμιλοι, οι βιομηχανικοί με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνεργαστούν σε όλους αυτούς τους μεγάλους ε, τομείς όπου υπάρχουν ακόμα προ δυνατότητες ανάπτυξης. Και ξέρουμε ότι στα τελευταία μεγάλα έξι προγράμματα οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι, μεγάλες, οι μεγάλοι όμιλοι ουσιαστικά μπόρεσαν να πάρουν τις περισσότερες δυνατότητες γιατί δεν μπορούσαμε καν να δούμε τις προδιαγραφές στην αρχή. Πώς μπορούμε εμείς να προτείνουμε κάτι το ε, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες ενός προγράμματος αν δεν έχουμε καν τη δυνατότητα να γνωρίζουμε εγκαίρως προς τα που πάει ένα πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε ότι δημοσιεύεται, ανακοινώνεται επίσημα κάτι, οι πρώτοι που μπορούν να το δουν και να υποβάλουν προτάσεις είναι οι μεγάλοι όμιλοι και εμείς πιστεύουμε ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, αν μας δείξετε προς τα που πρέπει να πάμε, μπορούμε να προσαρμοστούμε πολύ καλύτερα. Δώστε μας σωστά μηνύματα, παρουσιάστε μας σωστά τα προγράμματα και μη μας δίνετε μόνο ένα μικρό φωτάκι όταν έχει ήδη προχωρήσει, έχει ήδη εντοπιστεί από τους μεγάλους ομίλους το πρόγραμμα, έχουν ήδη υποβάλει τις προτάσεις τους. Από τις μεγάλες μέχρι τις μεσαίες, τις μικρές επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να ε, συμμετάσχουν. Επίσης μας ρωτήσατε αν εμείς μπορούμε εύκολα να συνεργαστούμε με μεγάλους ομίλους. Βεβαίως, δεν υπάρχει εδώ ανταγωνισμός. Εμείς αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξέρουμε οι μεγάλοι όμιλοι προς τα που παν, τι πληροφορίες έχουν, έτσι ώστε και εμείς να συγχρονιστούμε, να προσαρμοστούμε. Τους μεγάλους βεβαίως και τους χρειαζόμαστε. Είτε πρόκειται για μεγάλα προγράμματα στον διαστημικό τομέα, στον τομέα των ε, δορυφόρων, είτε πρόκειται για το πρόγραμμα ανάπτυξης του Airbus. Επαναλαμβάνω, οι μεγάλοι όμιλοι θα πρέπει απλώς να μας αφήσουν και εμείς να διαβλέψουμε προς τα που υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης και σαφώς μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους και να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες με βεβαίως τις αρχές του θεμητού ανταγωνισμού. Ο καθένας στο δικό του επίπεδο, στη δική του εμβέλεια μπορεί να συμμετάσχει. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι βεβαίως να ξέρουμε ποιο θα είναι το ποσοστό που θέλετε να διαθέσετε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην λέτε μονίμως ναι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται δουλειά, άρα θα σας δώσουμε ε, ένα μικρό ποσοστό. Όχι. Αυτό που θέλουμε είναι να συμμετέχουμε εκεί που μπορούμε να προσθέσουμε κάτι, εκεί που προσφέρουμε προς τη θέμενη αξία, εκεί που είμαστε ανταγωνιστικοί και ισχυροί. Υπάρχουν δυνατότητες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουν και οι μεγάλοι όμιλοι αλλά και οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις πώς μπορούν να συνεργαστούν. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι που επειδή είναι εμπιστευτικός ο χαρακτήρας των προγραμμάτων αυτών, πολλές φορές δεν είναι εύκολο να δημοσιευθεί και να ανακοινωθεί εγκαίρως. Βεβαίως έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες στην καινοτομία, οι συνεργασίες είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και στον τομέα των νέων τεχνολογιών, αλλά οπωσδήποτε σήμερα υπάρχουν ε, επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό, δεν μπορούν να επιβιώσουν εάν δεν ε, υπάρξει άμεση στήριξη. Βεβαίως ο τομέας ε, ο αμυντικός προσφέρει δυνατότητες, εμείς περιμένουμε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες για να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, η ΑΕΣΔ μπορούν να συνεργαστούν έτσι ώστε να βρεθούν αυτές οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν. Επαναλαμβάνω ότι εμείς πολλές φορές δεν έχουμε τη δυνατότητα να περιμένουμε πάρα πολύ για χρηματοδότηση. Και αν υπάρχει υπερβολικά μεγάλη ε, διαδικασία, γραφειοκρατία και αναμονή, κινδυνεύουμε να μην μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Η συνεργασία, αν θέλετε, θα πρέπει να επιτρέπει στις δικές μας μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το αποσαφηνίσω είναι ότι έχουμε δραστηριότητα και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και εμείς να συμμετάσχουμε σε προγράμματα ερευνητικά ή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ότι τα τελευταία 7-10 χρόνια η ASD υποβάλλει προτάσεις ε, για το πρόγραμμα πλαίσιο. Σε κάποια από αυτά έχουμε πετύχει, έχουμε στηριχθεί, έχουμε χρηματοδοτηθεί και πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές συνεργαζόμαστε με εταιρείες άλλων ευρωπαϊκών ε, κρατών, με ανταγωνιστές μας πολλές φορές και πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία και μεταξύ ε, μεγάλων και μεσαίων ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει προχωρήσει με επιτυχία, αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχει ένα οργανισμός ή μια επιχείρηση ήδη δραστηριοποιηθεί, να έχει τεχνογνωσία, να έχει αποτελέσματα σε ένα τομέα έτσι ώστε να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα συνεργασίας. Οι δικές μας δυνατότητες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βοηθήσουν την Ευρώπη να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της ε, στο ε, διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή, ο κύριος Γκάλερ. Ναι, επανέρχομαι στο θέμα της πιστοποίησης. Είπατε ότι είσαστε υπέρ της πιστοποίησης αλλά θα προτιμούσατε να υπάρχει ένα πιστοποιητικό που να ισχύει για όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε να μην αναγκάζεστε κάθε φορά να ανταποκρίνεστε στις προδιαγραφές της κάθε χώρας. Τι κάνετε σήμερα. Ένα προϊόν παράγεται, αναπτύσσεται, ολοκληρώνεται και κατόπιν ζητάτε την πιστοποίηση για τις ε, στρατιωτικές χρήσεις, για την μη στρατιωτική χρήση, για την κάθε χρήση υπάρχουν διαφορετικές διαγραφές, άρα διαφορετική πιστοποίηση. Επίσης σήμερα υπάρχουν διαφορετικά πιστοποιητικά σε όλες τις χώρες. Το ερώτημα λοιπόν αυτό πρέπει να στραφεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε αυτές τις διαδικασίες έτσι ώστε πρώτον να γίνονται μία φορά οι αιτήσει για πιστοποίηση έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε και χρόνο και χρήμα. Θέλετε να απαντήσετε αυτή την ερώτηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. All, the panelists, okay. Well, I guess so two, two, two minutes each, yes, I propose. Mr. Goss was also had something important to say. But what we say in the communication is simply... Όπως λέει η ανακοίνωση, εμείς βλέπουμε που είναι το πρόβλημα. Η πιστοποίηση ενός προϊόντος σε 27 χώρες είναι χρονοβόρα και χρηματοβόρα φυσικά. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες που έχουμε, σαν ε, ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία πιστοποιεί τα πολιτικά αεροσκάφη, είναι να το αντιμετωπίσουμε με πιο ευρωπαϊκό τρόπο. Βέβαια το θέμα ανήκει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών να το αποφασίσουν αυτό. Μέχρι τώρα έχει γίνει μια κάποια προσπάθεια. Εμείς προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε την αντίστοιχη διαδικασία στην πολιτική αεροπορία με ευρύτερο τρόπο και πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός αυτός στο μέλλον θα μπορέσει να λειτουργήσει. Εάν δείτε τι συμβαίνει στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Ε, θα δείτε ότι βρισκόμαστε σήμερα στην κατάσταση που βρισκόμασταν στην πολιτική αεροπορία πριν 20 χρόνια. Μπορούμε λοιπόν να ε, θέσουμε στόχους, να σεβαστούμε φυσικά τις εθνικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις και να εκμεταλλευτούμε την προσπάθεια η οποία έχει γίνει μέχρι τώρα. Να προσθέσω σε αυτό που είπε ο κύριος Τουκόσκι. Ε, είμαστε δραστήριοι στον τομέα αυτό γιατί υπάρχουν δυνατότητες ε, πολλές από την ενιαία ή πιο ολοκληρωμένη εναρμονισμένη διαδικασία πιστοποίησης. Όπως είπατε ότι έγινε και στην περίπτωση του Α400M, τώρα τα πράγματα προσπαθούμε να τα κάνουμε καλύτερα γιατί κάθε στρατιωτικό αντικείμενο, όχι μόνο ε, ε, αεροσκάφη αλλά και τεφαρακισμένα οχήματα ή οτιδήποτε άλλο πάντα η διαδικασία πιστοποίησης είναι μια αυστηρά εθνική μέχρι τώρα διαδικασία. Προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε εκ των υστέρων. Δεν είμαστε πάντα 27-28 χώρες σε τέτοιου είδους, αλλά υπάρχει μια ομάδα χωρών η οποία θέλει να συνεργαστεί με την ΕΑΖΑ σαν παράδειγμα εμείς σαν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία έχουμε μια συμφωνία συνεργασίας για να ασχοληθούμε και με τα στρατιωτικά θέματα σε συνεργασία με την ΕΑΖΑ για τα κράτη-μέλη. Για μας, εκ μέρους της ΑΕΣΔ, βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες εργασίας που ασχολούνται με το θέμα της πιστοποίησης, της ε, εναρμόνισης ε, των προδιαγραφών και βεβαίως εδώ υπάρχουν εκπρόσωποι από τις ε, εθνικές βιομηχανίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει κάποια στιγμή μια ενιαία διαδικασία. Βεβαίως το θέμα του εξοπλιστικού τομέα και της πιστοποίησης δεν είναι εύκολο να υπάρξει ενιαία διαδικασία στον τομέα αυτό. Απ' την άλλη μεριά, και αυτή είναι η προσωπική μου βεβαίως άποψη, υπάρχει και το θέμα των χρονοβόρων διαδικασιών, αλλά και το πώς θα δείξουμε ότι πραγματικά κοιτούμε το οικονομικό κομμάτι οι στρατιωτικές, ε, αν θέλετε, παραγωγές εξοπλισμών, οι στρατιωτικές διαδικασίες ε, δεν μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις απαιτήσεις χρόνου και εξοικονόμησης ε, ενός προϊόντος που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για αμυντικούς λόγους ενιαίες λοιπόν διαδικασίες, τα κοινά πρότυπα, η πιστοποίηση. Είδατε παραδείγματος χάρη τι έγινε με την οδηγία REACH. Προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να υλοποιηθούν. Τι θα γίνει με τις διαφορετικές προδιαγραφές και παραδόσεις που ισχύουν στις εθνικές αγορές. Για να σας πω λοιπόν καταρχήν την άποψή μας, εμείς στην ΑΕΣΔ έχουμε ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχοληθεί με το θέμα αυτό, το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό και προσπαθούμε τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ενιοποιήσουμε λίγο τα κριτήρια, τον τρόπο που εργαζόμαστε και τις απαιτήσει για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το πάνελ, σε αυτή την ακρόαση για τα σχόλιά σας. Η Υποεπιτροπή θα συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στα διάφορα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπορώ λοιπόν απλώς να σας ενημερώσω ότι στις 27 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή στις 9.30 το πρωί εδώ στις Βρυξέλλες τέλος της συνεδρίας και σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την παρουσία σας εδώ.